ενθαρρύνετε τις χώρες σας να προωθήσουν το νούμερο αυτό. Ευχαριστώ. Αδελφοί, η συζήτηση γύρω από την προφορική ερώτηση έληξε και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Κάμερβερτ για τη συνδεδεμένη τηλεόραση και ήθελα να παρακαλέσω την ε, εισηγήτρια να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω πρώτα πρώτο σκιώδη εισηγητή και την σκιώδη εισηγήτρια για τη βοήθειά τους. Είναι επίκαιρη η έκθεση αυτή ε, για την Ευρώπη διότι σήμερα ε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, ορίσουμε συγκεκριμένους κανόνες ούτως όταν η κατάσταση ψηφιακής αγοράς είναι αυτή που λέγαμε το πρωί υπάρχουν ε, πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τις μεν τεχνολογίες που ως αντίπαλες των δε. Αυτό είναι λάθος. Ε, στις περιστάσεις που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να διαλέξουμε τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης, επικοινωνίας δεν είναι, εμπορεύματα αλλά είναι και κοινωνικά αγαθά και ε, βεβαίως η αγορά ε, ε, ξαφνικά δέχεται νέους παίκτες αυτούς που φτιάχνουν τις πλατφόρμες, αυτούς που φτιάχνουν ε, καινούργια, ε, ε εφαρμογές. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τελικά ορίζουν και το περιεχόμενο το οποίο επικοινωνείται στον ε, χρήστη. Ε, εμείς ε, που είμαστε πέρα από τις εταιρείες αυτές θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε αφήσουμε μόνο τις εταιρείες να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις ή έχουμε μιλήσει για την, ε, τις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα για το ότι ο τομέας μπορεί να αυτορυθμιστεί και τα λοιπά από εκεί και πέρα ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν καταχρήσεις αλλά δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην καταγγελία εξόφθαλμων καταχρήσεων και να αφήνουμε ας πούμε τη διαφήμιση να διαφημίζει οτιδήποτε θέλει. Είναι ε, θα πρέπει να προωθήσουμε, ε, να καλύψουμε αν θέλετε κοινωνικές ανάγκες και ε, γενικά ενδιαφέροντα τα οποία μπορεί να μην είναι εμπορικά. Δεν είναι δυνατόν μόνο ο κατασκευαστής της πλατφόρμας ή των διαφόρων εξοπλισμών να αποφασίζει για το περιεχόμενο. Θα πρέπει να το αποφασίσουμε εμείς. Θα πρέπει επίσης να, να εξασφαλίσουμε ότι οι εφαρμογές και οι πρόσβαση και οι εφαρμογές είναι απλές. Θα πρέπει να μέσω των ρυθμιστικών υπηρεσιών αρχών να φροντίσουν να φροντίσουμε εμείς να ε, υπάρχει και συνένεση του αυτού που παρακολουθεί, που χρησιμοποιεί τις ε, καινούργιες τηλεοράσεις. Μέχρι στιγμής οι κανόνες που υπάρχουν αφορούν μοναχά γραμμική επικοινωνία. Οι μη γραμμικές επικοινωνίες έχουν ε, αφαιθεί πιο ελεύθερες. Γι' αυτό πρέπει να παρέμβουμε και να και φροντίσουμε οι νέες τεχνολογίες να ακολουθούν και αυτές κάποιο κανόνα. Από εκεί και πέρα το τι βλέπει ο κάθε ε, ακροατής, ο κάθε χρήστης τηλεόρασης είναι δικό του θέμα το να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τον χρήστη με συγκεκριμένα δεδομένα είναι λάθος και είναι και επικίνδυνο και άπτεται των βασικών δικαιωμάτων του ακροατή ο οποίος πρέπει να παραμείνει ανώνυμος. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και πιστεύω ότι στο μέλλον θα κάνουμε πολλές πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Κάμερβερτ, περνάμε στην ε, διαδικασία Catch the Eye. Θέλω να δώσω πρώτα το λόγο στην συνάδελφο Φερχάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση της ε, Πέτρα Κάμερα νομίζω τονίζει ένα φαινόμενο γιατί πλέον βλέπουμε πως τα δεδομένα χάνονται στο ίντερνετ. Οι έξυπνες τηλεοράσεις αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή σύγκλησης των έξυπνων νέσων και έχουμε τη σύγκληση της κλασικής ραδιοτηλεόρασης με τις δυνατότητες προσφέρει το διαδίκτυο. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για τον οπτικοακουστικό τομέα, γιατί βεβαίως η κλασική τηλεόραση έχει πολύ πιο αυστηρή ρύθμιση σε αντίθεση με το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και όμως βρίσκονται αυτά στα, ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη, οπότε θα μπορούσαμε νομίζω να το ρυθμίσουμε λαμβάνοντα υπόψη και την κοινωνική σημασία της ραδιοτηλεόρασης. Ε, θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε αυτό το ζήτημα και στο μέλλον. Με την έκθεση αυτή γίνεται ένα πρώτο βήμα προς σωστή κατεύθυνση και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Το πολύ, ο συνάδελφος Βέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού. Η κυρία Κάμερεβερτα ασχολήθηκε με ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Η τηλεόραση έχει μεγάλη ισχύ στην ε, κοινωνία και η φυστάμενη οπτικοακουστική οδηγία καλύπτει μόνο την τηλεόραση αλλά πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον θα εμφανιστούν νέες τεχνολογίες ε, που θα συνδυάζουν τηλεόραση και άλλα μέσα και θα έχουν όλο και μεγαλύτερη εξουσία οι κατασκευαστές αυτών των ε, συσκευών. Γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε τώρα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τη λεγόμενη συνδεδεμένη τηλεόραση, να μιλήσουμε για την διαθεσιμότητα, προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά. Και βεβαίως να είναι συμβατές οι συσκευές. Χίρς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Ε, κύριε Επιτροπέ. Φαντάζεστε βεβαίω πως εμείς ε, ως φιλελεύθεροι απορρίπτουμε αυτή την έκθεση. Πρόκειται περί λογοκρισία. Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει, δεν αναφέρεται ρητό στην έκθεση. Ναι, ναι, ναι κυρία Κάμερεβερτ. Δεν μπορεί να ρυθμίζουμε τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμίζουμε από την πολιτική το τι θα βλέπει ο κάθε ένα στην τηλεόρασή του. Δεν μπορεί να λέμε αυτό είναι καλό, αυτό είναι άσχημο, αυτό μπορεί να το βρει εύκολα και γρήγορα, όλα τα άλλα, ό,τι δεν μας αρέσει δηλαδή, να το κρύψουμε. Είναι το πρώτο βήμα προς τη λογοκρισία αυτό. Αυτό δεν το θέλουμε ως φιλελεύθεροι. Πρέπει ε, να υπάρχει ποικιλομορφία και στο μέλλον και μέσω της... Ε, ραδιοτηλεόρασης. Εσείς μας λέτε πως απειλείται η γνώση μέσω της ε, ποικιλομορφίας. Δεν είναι δυνατόν. Ήρθε η συνάδελφος Μακλάρκιν. Well, connected TV is an exciting innovation. Η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι μια εντυπωσιακή καινοτομία. Τέτοιες πλατφόρμες υπάρχουν ήδη σε πολλά σπίτια, αλλά είμαστε ακόμα στις αρχές αυτής της επανάστασης όσον αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού. Η έκθεση αυτή τονίζει τις προκλήσεις όσον αφορά το πλουραλισμό των μέσων, τις διαφημίσεις για τους νέους και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο θεμητός ανταγωνισμός ανάμεσα στους προμηθευτε... ευρωπαίους προμηθευτές περιεχομένου και τις μεγάλες πλατφόρμες που δεν υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανήλικους ε, με μέτρα που δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή για το ίντερνετ. Ε, γι' αυτό και ζητάμε από την Επιτροπή να εξετάσει ένα κατάλληλο, ε, να εξασφαλίσει μάλλον ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε το περιεχόμενο να είναι ποιοτικό, είτε παρέχεται από μια ε, διεθνή πλατφόρμα είτε από μια ευρωπαϊκή. Ε, δεν μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι μια πολυτέλεια την οποία θα χαίρουν μόνο οι πολίτε σε αστικέ περιοχέ όπου η ταχύτητα του Ιντερνετ είναι πολύ γρήγορη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούμε συνδεδεμένη τηλεόραση. Σημαίνει μια ευρυδική τηλεόραση παραδοσιακή και διαδικτυακή. Α, αν θέλουμε αυτή τη τηλεόραση να επιτύχει θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι γίνεται. Η παραδοσιακή τηλεόραση είναι πλέον ιστορία. Ήδη υπάρχουν συσκευές οι οποίες αγοράζονται, πουλούνται και αγοράζονται και οι οποίες ε, περιλαμβάνουν και το διαδίκτυο υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται και με αυτή την έννοια οι καινούργιες αυτές οι βρυδικές συσκευές είναι μια πρόκληση για η διαφήμιση και η προστασία των ανηλίκων εξασφαλίζεται με αυτές τις νέες συσκευές όμως αυτό βέβαια σχετίζεται με το τι θα κάνουν οι εθνικές αρχές για τη νέα τεχνολογία Μπορείς Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια από την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων για την έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή γιατί πραγματικά η αγορά για την οποία συζητούμε ε, αλλάζει. Έχουμε καλλιδιακή τηλεόραση, έχουμε ψηφιακή τηλεόραση, έχουμε το διαδίκτυο και σύγκληση όλων αυτών των μέσων δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Ε, θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας ε, από ορισμένες εκπομπές στην τηλεόραση, από τη διαφήμιση και τα λοιπά. Το βεβαίως ε, ο χρήστης πρέπει να μπορεί να συνενεί ή όχι. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Επίσης οι βαρύκοοι ή οι άνθρωποι με αναπηρίες θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες αυτές τεχνολογίες και όσον αφορά τους κανόνες θα πρέπει πραγματικά να υπάρχουν και εδώ οι κανόνες που υπάρχουν για τις γραμμικές υπηρεσίες. Είναι πολύ καλή η συζήτηση που γίνεται εδώ. Ο Επίτροπος Χάν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευρυδική τηλεόραση. Αναφέρονται πολλά ζητήματα και φαίνεται με, ακριβώς πόσο πολύπλοκος είναι ο οπτικοακουστικός τομέας. πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα ε, έγγραφο επί του οποίου θα βασιστεί και η δημόσια διαβούλευση που γίνεται για τον οπτικό-ακουστικό τομέα. Γιατί πραγματικά είναι η νέα κατάσταση δημιουργεί και ευκαιρίες και προκλήσεις που άπτονται των βασικών αξιών και αρχών της Ένωσης η έκθεση της κυρίας Κάμερβερτ θα χρησιμοποιηθεί και αυτή πέρα από την πράσινη βίβλο για τη διαβούλευση που κάνουμε και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και τη σημασία του, των ρυθμιστικών αρχών και του, του ρυθμιστικού συστήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύγκληση στον οπτικοακουστικό τομέα. Ξέρουμε, έχουμε την οδήγηση τη, μια οδηγία σχετική. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλο, πολλές και διαφορετικές απόψεις. Πολλοί πιστεύουν ότι η οδηγία που εγκρίθηκε λειτουργεί καλά. Α, και αναφέρθηκε επίσης το θέμα της αυτορύθμισης του κλάδου. Όλα αυτά αναφέρονται στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι, ότι ε, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία για τον οπτικοακουστικό τομέα μετά το τέλος της διαβούλευσης. Θα το δούμε. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013. Ε, προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάληψη κατόπιν αυτού πρωτοβουλειών και μέτρων. Η Κομισιόν έχει σαν στόχο να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη με σύγχρονη όμως προστασία των αρχών και της ε, πυκλομορφίας. Η θα διεξαχθεί ε, σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Πέντε λεπτά διακοπή για να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ.